Επιτροπή για τις ε, ε, κυρώσεις που έχει επιβάλει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο, και επηρεάζουν τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράν. Περιμένουμε δύο λεπτά. Ναι, περιμένουμε τον κύριο Λάγκ. Ε, Σα ζητώ υπομονή λιγόλεπτη και αν ε, όντω ε, δεν θα έρθει θα συνεχίσουμε με την κυρία Μπιενκόφσκα. Ευχαριστώ για την πρότασή σας. Nous allons pouvoir reprendre la séance. Θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τώρα, κατέθεσε ο κύριος Λάνια. Του δίνουμε ένα λεπτό ε, για να ε, πάρετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε. Είχα την πληροφορία ότι θα αρχίζαμε στις 19 και 16 τη συζήτηση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, όντως η προφορική ερώτηση αναφέρεται στις επιπτώσεις των κυρώσεων των Ενωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν και τις επιπτώσεις δηλαδή που έχουν οι κυρώσεις αυτές σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Έχουμε αυτό, αυτή τη συμφωνία για τα πυρηνικά που επετεύχθη με το Ιράν και συνεπέφερε την άρση των κυρώσεων. Καταρχήν θετικό προωθείται η συμφωνία αυτή με το Ιράν και ενισχύεται και η διαδικασία οικονομικής ανοικοδόμησης της χώρας αυτής. Ωστόσο, υπάρχουμε το πρόβλημα ότι πολλές αμερικανικές κυρώσεις είχαν ήδη επιβληθεί από το 1979, πριν δηλαδή από την πυρηνική προσπάθεια του Ιράν. Ιράν. Και αυτές δεν έχουν αρθεί. Έχουν λοιπόν μια εξοεδαφική επίπτωση και σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Με την έννοια αυτή ε, είναι σωστό να εγγύψει κανείς το ερώτημα ε, πώς, πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Διότι αποδεδειγμένα υπήρξαν επιπτώσεις σε ορισμένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αλλά ορισμένες από αυτές μετά από έντονες συζητήσεις με τις Αμερικανικές αρχές έλαβαν κάποια εξαίρεση. Παρ' όλα αυτά, διαπιστώνεται μια άνηση μεταχείριση μεταξύ Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει σαφήνεια, να ξεκαθαριστεί το θέμα των εξοεδαφικών επιπτώσεων των κυρώσεων. Και ιδίως αναφέρομαι στον τραπεζικό τομέα την πρόσβαση δηλαδή σε χρηματοδοτήσεις, δεν είναι δυνατόν να αποκλείονται ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την ε, λογική χρηματοδότηση των έργων που αναλαμβάνουν. Πρέπει όλοι να μπορούν να υποφεληθούν από τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται για δουλειές με το Ιράν και ιδίως για την σταθεροποίηση της περιοχής αυτής και για την ανάπτυξη της Ιρανικής κοινωνίας, κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Γι' αυτό ως Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου διατυπώσαμε την προφορική αυτή ερώτηση πώς δηλαδή κρίνει την κατάσταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς θα την αντιμετωπίσει με μέτρα, με την λήψη μέτρων για να διασφαλίσει την εφαρμογή των, την υλοποίηση δηλαδή των υπεσχημένων να ξεκαθαρίσει απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείε ότι αυτές οι εξωεδαφικές κυρώσεις δεν επιτρέπεται να έχουν επιπτώσεις σε ευρωπαϊκές εταιρείε. Το ερώτημα λοιπόν είναι πρώτα αν έχετε συζητήσει με τους Αμερικανούς και τι σας απάντησαν. Τέλος, η ερώτησή μου είναι πώς θα μπορέσετε ή πώς θα θελήσετε να διασφαλίσετε τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μέσα στα πλαίσια αυτά. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ και πάλι συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Λάγκε και η κυρία Μπιέν Κόψκα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο κύριε. Σας ευχαριστώ. Ε, πέντε ε, μήνες μετά την άριστον των οικονομικών ε, κυρώσεων, με, μετά την εφαρμογή από το Ιράν των υποχρεώσεων του ε, βάσει της Περνικής ε, Συμφωνίας ε, γίνεται αναθεώρηση των σχέσεων και των επιπτώσεων που υπάρχουν για τις οικονομικές σχέσεις με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να τονίσω πως ο η απαιτούμενη προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την επιτυχία της ε, συμφωνίας ε, είναι ε, να εξασφαλίσουμε τα οικονομικά ωφέλη για όλες, τις, για πλευρές. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι όταν θα επισκεφθεί η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος και 7 άλλοι επίτροποι το Ιράν θα πάω και εγώ εξάλλου στην Τεχεράνη τον Πήγαμε μάλλον στη Χεράνη τον Απρίλιο και διαπιστώσαμε ε, ότι ε, υπάρχει ε, σοβαρό ενδιαφέρον για την σωστή εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. υπάρχει ο συντενιστικός ρόλος της ΥΠΑ εκπροσώπου ε, και βάσει αυτού υπάρχει συστηματική υποπτία της εφαρμογής της ε, συμφωνίας. Ε, όπως συμφωνήσαμε στο σχέδιο δράσης έχουν αρθεί οι κυρώσεις, έχουν εκδοθεί συστάσεις και άρα επικρατεί σαφήνεια σε σχέση με τη στάση μας ως προς αυτά τα ζητήματα. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται διαφάνεια και σαφήνεια για το ιδιωτικό τομέα γιατί πρέπει να επιστρέψουν οι επενδυτές στο Ιράν. Ε, Α είμαστε ξεκάθαροι, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και άλλε προκλήσει. Υπάρχουν τα χρηματοπιστωτικά και τραπεζικά ζητήματα και θα πρέπει να υποτιμήσουμε πόσο μεγάλε είναι οι δυσκολίε. Όμω θα πρέπει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα, διότι πάνω από 10 χρόνια είχε απομονωθεί οικονομικά το Ιράν. Οι τράπεζε είχαν αποκοπεί ε, για αυτή τη δεκαετία από το διεθνέ χρηματοπιστωτικό σύστημα και ξέραμε ανέκαθεν ότι η πλήρη ενσωμάτωσή του Ιράν στην παγκόσμια οικονομία δεν θα συμβεί νυχθημερών, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Θα στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα. Ε, λαμβάνεται υπόψη αυτό από πολλά τραπεζικά ιδρύματα ανά τον κόσμο και ε, ε, είναι μεγάλο το πεδίο των των επιπτώσεων των οικονομικών ακυρώσεων ε, της ΕΠΑ. Επίσης υπάρχουν οι έλεγχοι σε σχέση με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και αυτές έχουν επιπτώσεις στις οικονομικές σχέσεις και στα δύο μέτωπα δραστηριοποιούμαστε και συστηματικά ε, έχουμε διαβουλεύσεις με την Washington από τις 16 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και ε, δύο φορές επικαιροποιήθηκαν οι συστάσεις, δημοσιεύθηκαν νέες συχνές ερωτήσεις για τους επιχειρήσεις επιχειρηματίες, ούτως ώστε οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λειτουργούν σε ένα σαφές περιβάλλον ε, και καλέσαμε επίσης ε, τον ε, προϊστάμενο του Γραφείου των ε, Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχειών ε, να ενημερώσει τους υπουργούς μας και να απευθύνει έκκληση προς τους ιδιώτες επιχειρηματίες. Στις Βρυξέλλες θα διοργανώσουμε και συμπόσιο για την άζη των κυρώσεων για τους φορείς της επιχειρηματικής κοινότητα με εμπειρογνώμενος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη ΣΥΠΑ. Επίσης, διπουργική συνάντηση στις 19 Μαΐου με τους υπουργούς εξωτερικών της Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και ΙΠΑ και από εκεί προέκυψε μια κοινή δήλωση ε, για ε, τις επιχειρηματικές σχέσεις με το Ιράν μετά την άρση των κυρώσεων. Ήταν ένα σαφές μήνυμα προς τους επιχειρηματίες τους ώστε να αναθερμάνουν τι σχέσεις τους με αυτή τη χώρα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες ε, των ΗΠΑ να προσφέρουν μια σαφή εικόνα σε σχέση με την άρση των πρωτογενών κυρώσεων των ΗΠΑ και των εκκλήσεων που ευθύνουν προς τον τραπεζικό τομέα συγκεκριμένα. Είναι επίση σημαντικό όμω όμω ε, σε κανονιστικό και επιχειρηματικό επίπεδο και το Ιράν ε, να αναλάβει τα απαιτούμενα μέτρα. Ανησυχούν επιχειρήσει και διάφορα ζητήματα για την νομοθεσία, για την ε, νομοποίηση στον παράνομων δραστηριότητε, για σχέση με την νομοθεσία κατά της χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Πρέπει να κάνει περισσότερα το Ιράν. Επίσης, ε, σε προτεραιότητα θα πρέπει να αναδειχθούν οι συστάσεις ε, της ειδική Task Force. Ε, το Ιράν προσφέρει μια βάση συνεργασίας και συνεργάζεται μαζί μας. Παρόλες αυτέ τι μεγάλες προκλήσεις, το αποτέλεσμα του προγράμματός μας είναι θετικό. 27% αύξηση των επιχειρηματικών σχέσεων στο πρώτο τετράμινο του 2016, αν το συγκρίνουμε με το 2015 33 ε, ε, τράπεζες του Ιράν ε, επανασυνδέθηκαν με το SWIFT μέχρι στιγμής και 200 μικρομεσές διεθνείς τράπεζες και ευρωπαϊκές άρχισαν να αποκαθιστούν τις σχέσεις τους με τις τράπεζες του Ιράν και νιώθουν μεγαλύτερη άνεση διότι στην πράξη αντιλαμβάνονται πώς μπορούν πλέον να λειτουργήσουν σε συνεργασία με το Ιράν. Τον Οκτώβρη έχουμε προγραμματίσει σε μια νέα αποστολή οικονομικών φορέων στο Ιράν με τους εκπροσώπους Ευρωπαίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων διότι έτσι μπορούμε να προωθήσουμε τις επιχειρηματικές σχέσεις και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις ασφαλιστικές εταιρείες ε, διότι αυτό θα καθησυχάσει περισσότερο ε, τους ιδιώτες επενδυτές. Όλα αυτά τα ζητήματα ε, ε, αποτελούν από κοινού την περίπλοκη πραγματικότητα που ζούμε στις σχέσεις μας με το Ιράν. Φυσικά θα πρέπει να προσαρμοστεί η διεθνή κοινότητα στη νέα κατάσταση μετά την άρση των κυρώσεων. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τις τράπεζες ούτε τους επενδυτές να πάρουν κάποιες αποφάσεις παρόλα αυτά. Ε, αναλαμβάνουμε αυτή τη δέσμευση ούτως ώστε να μπορέσει και το Ιράν να αποκομίσει οικονομικά ωφέλη από αυτή την ε, συμφωνία. Συνεχίζουμε τη συνεργασία με τη ΣΥΠΑ, ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια ω προ του κανόνε που ισχύουν. Συνεχίζουμε τι εκκλήσεις προ την επιχειρηματική κοινότητα και την προσφορά τεχνική αρρωγή προ το χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό σύστημα του Ιράν. Αυτό είναι ο δρόμο που θα ακολουθήσουμε και στο μέλλον. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριο Μποστινάρου για τρία λεπτά από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε. Με χαρά πριν από ένα χρόνο είδα ότι υπήρξε ε, λύση μετά από τις δύσκολες και μακρές διαπραγματεύσεις ε, με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ρόλο κλειδί σε αυτή την επιτυχία και όπως είπα και τότε η συμφωνία θα πρέπει να ωφελήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ε, το κοινό πρόγραμμα δράσης που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο μπορεί να σημάνει σημαντική πρόοδο για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Όμως παραμένει εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμοστεί με καλή πίστη από όλα τα μέρη όσο γίνεται πιο σύντομα. Θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η συμφωνία ξεπερνά τις τεχνικές της, ε, τα τεχνικές της λεπτομέρειες και θα πρέπει να ε, τηρηθεί και από τον Ιρανικό λαό όταν θα ολοκληρωθεί. Ελπίζουμε ότι αυτό θα βελτιώσει τι συνθήκες διαβίωσής τους και είναι πολύ σημαντικό να, ε, να το εφαρμόσουμε σωστά και επιτυχώς γιατί αυτό θα μας επιτρέψει να δείξουμε τα ωφέλη της διπλωματίας και το πόσο αντιπαραγωγικός είναι ο, ο σκοταδισμός. Ε, παρόλα Αυτά έχουμε, έχουν οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει ακόμα μεγάλες δυσκολίες για πρόσβαση στην Ιρανική αγορά και αυτό οφείλεται στο ότι οι αμερικανικά κυρώσει ε, εξακολουθούν να ισχύουν και έχουν και εξοδευτικό αντίκτυπο. Γνωρίζουμε το σύνολο των ε, εταίρων, των Αμερικανών και τα προβλήματά τους ως για θέματα όπως η ασφάλεια και το θέμα της χρήσης βαλιστικών όπλων. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τις διόδους συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ ώστε να βρούμε ε, τρόπο αποκατάστασης και ίσως και μια προσωρινή λύση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες και να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα μαζί με τους Ιρανούς εταίρους μας την ασφάλεια και την νομική ασφάλεια ε, βεβαιότητα για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στο Ιράν. Τέλος, κυρία Επίτροπε, η Κομισιόν θα πρέπει να προωθήσει την υιοθέτηση ενός νέου μηχανισμού και μέτρων για να μειωθεί η εξάρτηση των ευρωπαϊκών εταιριών από τις αμερικανικές πιστώσεις και τα ασφαλιστικά ιδρύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαχαρντήλ μόλις έφτασε, οπότε του δίνω το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ. Já ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Επιτροπή μου, στην ΙΝΤΑ, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διάφορες χώρες και είναι πρόθυμοι να στηρίξουν κάθε είδους κυρώσεις κατά χωρών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, πιστεύω πως αυτό δεν ε, ισχύει για το Ιράν ε, και ότι η ουσία αυτής της θεοκρατικής δικτορίας ε, υποτιμάται από πλευράς μας. Υπάρχει μια μετακίνηση στην κοινωνία που ακόμα δεν έχει, γίνει, δεν έχει αντικατοπιστεί στις κυβερνητικές δομές. Είναι μια θεοκρατική ε, μαζί με τη Ρωσία, τον Ασάντ και το Σχεσμπολά ε, είναι κατά της, ε, του δυτικού πολιτισμού. Ε, είναι μια χώρα που ποτέ δεν έχει εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες, γι' αυτό και συστήνω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις σχέσεις με το Ιράν. Ευχαριστώ, Σχάκε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Συζητάμε για να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για τις ευρωπαϊκές εταιρείε που ε, προσβλέπουν στο εμπόριο με το Ιράν μετά από την άρση των κυρώσεων, μετά από τη νέα συμφωνία. Όμως συνεχίζονται οι αμερικανικές κυρώσει για την παραβίαση ε, ε, των, ανθρωπιστικών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οδήγησαν σε αβεβαιότητα όμως για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ως αποτέλεσμα της του εξοδευτικού αντικτύπου Γι' αυτό και πολλές εταιρείες ε, ε, κάνουν πίσω. Χρειάζεται εξασφάλιση για το ότι οι τράπεζες θα, ας πούμε, θα είναι βέβαιες ότι οι υπηρεσίες τους δεν θα ε, τιμωρηθούν ε, από τις ΙΠΑ εάν ε, λειτουργήσουν εκεί. Όχι μόνο τα πρόστιμα, αλλά και οι απαιτήσει θεώρησης εμποδίζουν την πρόσβαση στις ΣΥΠΑ αφού κανείς έχει επιχειρήσει στο Ιράν. Ο Υπουργό Εξωτερικών Κέρι ε, ήρθε σε επαφή με τι Ευρωπαϊκέ Τράπεζε. Το θέμα είναι η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση τι έχουν κάνει για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα με την Αμερικανική κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει σαφήνεια και νομική βεβαιότητα για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Και τι κάνατε σε σχέση με τι Ιρανικέ αρχέ για το γεγονό ότι υπάρχει, έχει μεγάλο ρόλο η επαναστατική φρουρά στην Ιρανική οικονομία και αυτό εμποδίζει την ανάδυση ενό πραγματικά ιδιωτικού τομέα και επίσης κινδυνεύει τα ωφέλη μετά από τη συμφωνία να ωφελήσουν τους λίγους και όχι τους πολλούς. Είναι βασικό για την ομάδα μας και για την Ένωση, για να είναι αποτελεσματική και αξιοπιστή, να ασκήσουμε τις δικές μας πολιτικές σε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ όταν χρειάζεται, όπως με επιτυχία το κάναμε στο να επανέλθει το Ιρών στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, αλλά πάντοτε ανεξάρτητη βασιζόμενοι στις δικές μας εκτιμήσεις και αποφάσεις για το ποια εξωτερική πολιτική εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά μας και πάνω απ' όλα τις αξίες μας. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό έχει τώρα το λόγο κ. Κούσο Περμούη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ακολουθεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ και πάλι ε, βλέπει να περιορίζονται οι δυνατότητες εξωτερικής πολιτικής και εμπορικής πολιτικής. Ε, οι κυρώσεις αμερικανικές επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Είναι κυρώσεις ενάντια στο διεθνές δίκαιο και επηρεάζουν και πάνω απ' όλα τον λαό του Ιράν. Όπως έγινε και με τις κυρώσεις ε, κατά το Ιράκ το 1990, όπου σύμφωνα με το ΙΕ κόστησαν πάνω από μισό εκατομμύριο παιδιά, ε, νεκρά παιδιά. Έχουμε ακόμα το εμπάργκο στο κατάργαστο πετρέλαιο, όμως οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να έχουν δυσκολίες για να λειτουργήσουν στο Ιράν ως επίπτωση των εξοδευτικών ε, της εξοδευτικού αντικτύπου των Αμερικανικών κυρώσεων. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να κατηγορηθούν ότι παραβαίνουν τις Αμερικανικές κυρώσεις. Πού βρίσκεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κυριαρχία. Σας ευχαριστώ. Τώρα δύο λεπτό κύριος Μπούχνερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να ε, οδηγήσουμε σε λήξη την δεκαετία απομόνωση του Ιράν. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο εάν θέλουμε να συμβάλλουμε στην βελτίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην μείωση της τρομοκρατίας που προέρχεται από την ε, Μέση Ανατολή. Η κοινωνία στο Ιράν χρειάζεται την άρση των κυρώσεων, διότι υπάρχει ανεργία εκεί. Εκεί ζουν πολλοί άνθρωποι κάτω από τα στάνταρτ που θεωρούμε αναγκαία. Αυτά θα γίνουν όμως δυνατά μόνο με την ανάπτυξη του εμπορίου, με την άρση των κυρώσεων. Γι' αυτό θεωρώ ότι για να αναχαιτιστεί και η τάση προς τρομοκρατία και ριζοσπαστικοποίηση στην ίδια την κοινωνία του Ιράν, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο στην χώρα αυτή. Δεν μας μένει και τίποτε άλλο από το να ενισχύσουμε την οικονομική συνεργασία με την χώρα αυτή, να άρουμε τις κυρώσεις, έστω και αν έχουν κάποια ιστορική αιτιολόγηση από τη σκοπιά των ΗΠΑ. Θεωρώ ότι παρόλη αυτή την ενδεχόμενη ιστορική αιτιολόγηση είναι απαράδεκτο ευρωπαϊκές και γερμανικές επιχειρήσεις να υποχρεωμένες να τηρούν τις αμερικανικές κυρώσεις αυτό αποτελεί ε, θεμελιώδη αντίφαση στην κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ. Κύριε Μπούχνερ, θα, θα δεχτείτε μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Φονζελίκα. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ. Νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσει την εξοεδαφική επίπτωση των Αμερικανικών κυρώσεων και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μπορούν να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες ε, να μπορούν και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες χωρίς να φοβούνται αμερικανικές ε, ποινές, κυρώσεις και πρόστιμα. Ο κ. Μπούχνερ, θεωρώ πράγματι ότι οι κυρώσεις αυτές πρέπει να διευκρινιστούν σε διαπραγματεύσεις βεβαίως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των Πολιτειών. Συμφωνώ απολύτως με αυτό. Μάλιστα, δύο λεπτά, η κυρία Μπεγκίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Η ερώτησή μου είναι ποιο αποφασίζει του κανόνε που ισχύουν για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε, εμεί ή η Washington, γιατί από τον Οκτώβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταδιακά ήρε τι κυρώσει και επέτρεψε στι ευρωπαϊκέ εταιρείε να εμπορευθούν με το Ιράν. Αλλά όχι το είπα, που ακόμα ισχύουν οι δικέ του κυρώσει και εκτό που απαγορεύουν τι δικέ του επιχειρήσει να εμπορευθούν εκεί, ε, ε, βάζουν ε, αλμυρά πρόστιμα στις ευρωπαϊκές εταιρείες που το κάνουν. Και αυτό γιατί η Αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι οποιοδήποτε κάνει συναλλαγές με αυτή τη χώρα αναγνωρίζει μέσω στην κυριαρχία της. Είναι προφανές ότι το Ιράν ακόμα έχει δρόμο να διανύσει όσον αφορά τη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά, αλλά εφόσον από τότε μάλλον που οι κυρώσεις δεν μπλοκάρουν πια το εμπόριο, οι ευρωπαϊκές εταιρείες θέλουν να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν λόγω του εμπάρκου στην Ιρανική αγορά και είναι γελίο οι εταιρείε μα να μπλοκάρονται από την Αμερικανική κυβέρνηση, ενώ οι ευρωπαϊκέ ε, κυβερνήσει το επιτρέπουν. Α, μια Ιταλική τράπεζα, μεγάλη ε, ε, Ιταλική τράπεζα ε, έλαβε πρόστιμο και μια ε, εταιρεία Ιταλική ε, ερευνήθηκε αλλά χωρίς τελικά να πάρει πρόστιμο. Θα πρέπει ίσως, το, μάλλον η διαδικασία για να πάρει κανείς εξαίρεση από αυτές τις κυρώσεις είναι μακρά. Ε, και δαπανηρή. Ε, όπως είπα, είναι ο δρόμος μακρύς προς τη δημοκρατία για το Ιράν, αλλά αυτός ο δρόμος περνά και από τη σταδιακή ένταξη στο διεθνές εμπορικό σύστημα και κυρίως αν η Ευρώπη αποφάσισε να δώσει τη ε, το πράσινο φω τη επενδύσεις στο Ιράν, τον τελευταίο λόγο σίγουρα δεν θα πρέπει να τον έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπορκέτσιο, ένα λεπτό. Πρόεδρε, την παραμονή τη ψηφοφορία για το Brexit που είναι αύριο, θα, ήταν, ε, θα περιμέναμε μια θέση πιο δυναμική από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον για αυτά τα θέματα, εφόσον πρόκειται για την περάσπιση των ευρωπαϊκών ε, εταιριών. όμω, δεν καταλάβαμε ούτε καν ποια είναι οι κυρώσει κατά του Ιράν που ήραν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν υπάρχει σαφήνεια στα λόγια σας ενώ από πλευράς του Ιράν επαναλαμβάνονται διάφορα στις ευρωπαϊκές ε, εταιρείες οι προσκλήσεις να μπουν σε αυτή την αγορά που είναι λέει καταπληκτική. Η Ιταλία ε, ε, έχει πάρει πολλά πρόστιμα από την Γένοβα. Ένα σωρό βαπόρια είναι έτοιμα γεμάτα να φύγουν ε, με εμπορεύματα, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να τονώσει την οικονομία μας. Είναι απίστευτο η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι τόσο αδύναμη και αβέβαιη απέναντι σε ένα τέτοιο πρόβλημα που θα έλεγα ότι είναι καταφανώς συνδεδεμένο με τα συμφέροντα των επιχειρήσεών μας και των εργαζομένων μας. Ε, το Κοινοβούλιο, αντίθετα από την Κομισιόν, είναι ενωμένο και θέλει να καταργηθούν αυτές οι κυρώσεις και να μην επηρεάζουν τις, τις, τις δικές μας επιχειρήσεις οι οργανισμοί ελέγχου των Αμερικανών. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Γκόλνης. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συζήτηση που γίνεται για τι επιπτώσει των κυρώσεων, τον είπε, για τι δραστηριότητε των ε, επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ιράν. Ε, πρώτα απ' όλα γιατί εγώ ίδιο ε, υπέβαλα γραπτό ερώτημα πριν από δύο μήνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό και περιμένω ακόμη την απάντηση. Αφήστε που φαίνεται τι τελευταίε ημέρε ότι οι Αμερικανικέ αρχέ έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση σε σχέση με τι δικέ του επιχειρήσει. Δηλαδή, η άρση των κυρώσεων είναι για τι αμερικανικέ επιχειρήσει όχι για τις δικέ μα ε, και εξακολουθεί να υφίσταται η απειλή για τι δικέ μα επιχειρήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κύριο Κέλλη ε, ε, λέει ότι μπορεί κάποιο να δραστηριοποιηθεί στο Ιράν. Μάλιστα, αλλά η Airbus παραδείγματο χάρη περιμένει εδώ και μήνες το πράσινο φω από την αρμόδια αρχή για να πουλήσουν τα αεροσκάφη για τα οποία έχουν συμφωνήσει ήδη από το Ιανουάριο. Επίση, υπάρχει ένα τεράστιο δυστεό το πρόστιμο, δισεκατομμύρια δολάρια, 9 δισεκατομμύρια για την BNP, την Γαλλική Τράπεζα ε, και αδιαφορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αδιαφορούν όλοι είναι σκάνδαλο, είμαστε πραγματικά υποτελεί σε σχέση με την Ουάσιγκτον. Ε, ε, ευχαριστούμε κύριε Ζαφόλη. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η Συμφωνία της Βιέννης και η συνεπαγόμενη σταδιακή άρση των κυρώσεων θα πρέπει να θυμίσουμε ότι επέτρεψε από το 2005 μέχρι σήμερα να επιτρέψει την αύξηση κατά 70% των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράν. Πρόκειται για μια χώρα 80 εκατομμυρίων κατοίκων που αποτελεί τη μεγαλύτερη έλξη για τις διεθνείς ε, επενδύσεις μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Ε, μεταφορές, ε, καταπολέμηση της ε, ρήπανσης, κλιματικές αλλαγές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο δρόμος έχει χαραχθεί και τώρα όλοι οι φορείς που εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή η Ιράν, θα πρέπει μαζί να προχωρήσουν για να, και να βασιστούν σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και όχι μόνο στο σεβασμό των υπογεγραμμένων συμφωνιών. Από το Ιράν περιμένουμε μηνύματα ανοίγματο και αλλαγή με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ στο οικονομικό μέτωπο είναι απαραίτητο να δουλέψουμε κυρίως για το τραπεζικό σύστημα, γιατί μέχρι σήμερα δεν είναι διαφανές και επίσης υπό το φω των συστάσεων τη Task Force για την ε, ε, ε, χρηματοπιστωτική δράση, για να αποφύγουμε την ανακύκλωση χρήματος και να, αντιμετωπ... και καταπολεμήσουμε τους τρομοκράτες. Επίσης, ε, ε, ε, η ΕΠΑ μέχρι και τώρα εμποδίζουν τις επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε επιχείρηση δεν μπορεί ε, που συνεργάζεται έστω και κατά 2% με τη ΣΥΠΑ να κάνει δουλειές με το Ιράν. Ε, ε, ε περιορίζεται η ελευθερία δράσης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ζητάμε εντόνως λοιπόν από την Κομισιόν να μεταφέρει αυτό το μήνυμα προς τις Αμερικανικές αρχές. Είναι απαραίτητο τα ένα σωρό μνημόνια συνεννόησης που μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει δημόσιες και ιδιωτικέ επιχειρήσεις της Ευρώπης να μετατραπούν σε συμβάσεις και συγκεκριμένες δράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό. Μπάρεκοφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω αναλάβει το Ιράν στην Επιτροπή Ενέργειας το Ιράν πρέπει τώρα να υποφεληθεί από τις εξελίξεις αυτές. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προχωρούν σε αποκατάσταση ε, δεσμών με το Ιράν, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Αυτό χρειάζεται συνεργασία και με το Ιράν και με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και αυτό πρέπει να είναι το καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έρονται οι κυρώσεις. Πράγματι, όμως υπάρχουν πρόσθετες κυρώσεις από πλευρά των ΗΠΑ. Αυτό συμβαίνει λόγω της επιμονής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός κατέθεσε πρόταση για συνεργασία με το Ιράν. Από την άποψη αυτή θα μας υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι τα πράγματα καθυστερούν, χρονοτριβούμε. κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, δώσατε ή μάλλον θα δώσετε απάντηση σήμερα στην ερώτηση. Η απάντηση που δώσατε ήταν διπλή. Μιλήσατε για τις προσπάθειες που κάνετε και εσείς προσωπικά και οι συνάδελφοί σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέναντι στο Ιράν. Νομίζω ότι δώσατε πολλές πληροφορίες, είμαι βέβαιος ότι καταβάλατε σημαντικές προσπάθειες. Υπάρχει όμως ένα διπλό θεματολόγιο, διότι υπάρχει και το θεματολόγιο που αναφέρεται στην ποιότητα των δημοκρατικών εξελίξεων στο Ιράν, στα θεμελιώδη δικαιώματα κλπ. Από τη σκοπιά αυτή νομίζω ότι η απάντηση ήταν ικανοποιητική. Το άλλο τμήμα, έχω, για το άλλο θέμα έχω κάποιες δυσχέρειες για να είμαι ειλικρινής και εννοώ το τμήμα εκείνο που αφορά τις Ηνωμένε Πολιτείες. Απαντήσατε συντομότατα σε αυτό το μέρος της ερωτήσεως. Είπατε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος, υπάρχει κάποια πρόοδος ό,τι αφορά διευκρινήσεις που δίνονται και από τις δύο πλευρές και είμαι βέβαιος ότι έχετε δίκιο. Έχουμε όμως περιπτώσεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις. Είμαι Τσέχος. Υπάρχει μια περίπτωση και αυτή, ε, δηλαδή ε, πάρα πολύ έντονη, το Airbus και τα Boeing. Τα, η η εταιρεία Boeing άρχισε διαπραγματεύσει με το Ιράν πολύ αργότερα από την Airbus. Η Airbus αναμένει τώρα εδώ και ένα πεντάμινο την άδεια από, την, ε, από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ πρέπει να καταβάλλετε προσπάθειες οι οποίες να αποδώσουν αποτελέσματα. Πέστε μα αν μπορούμε και πώ να σα βοηθήσουμε. Αλλά πρέπει να αποδώσετε αποτέλεσματα. Ευχαριστώ κυρία Φων Στόρχη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Ιράν υπέγραψε την πυρηνική συμφωνία. Γι' αυτό Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε ήραν τι κυρώσει, όπω ακούσαμε, αλλά μόνο εν μέρη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εξακολουθούν ή μάλλον επαναλαμβάνουν το εμπόριο με το Ιράν. Έρχεται η General Electric και κάνει επιχειρήσει με το Ιράν. Όμω, όταν η Siemens πάει να κάνει το ίδιο, την απειλούν με κυρώσει οι Ηνωμένε Πολιτείε. Επομένω, το Ιράν στρέφεται στι Ηνωμένε Πολιτείε τότε για τι ε, ε, αυτές. Δεν είπατε, όπω προπαρτρίστηκε κάποιο άλλο προηγουμένω, γιατί δεν αντιδράτε. Το Exxon Mobile αγοράζει πετρέλαιο από, την, από το Ιράν και οποιαδήποτε άλλη αμερικανική επιχείρηση μπορεί να το κάνει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, αλλά και εμεί το ίδιο. Προτείνω λοιπόν αντί να επιβάλλουν κυρώσεις οι Ηνωμένες να τις άρουν. Ή απλώς αυτό που κάνουν είναι να, να υπερασπίζονται μάλλον την κυρίαρχη θέση τους. Ευχαριστώ. Κύριε Μπερτό, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Ιράν έδωσε όλες τις απαραίτητες εγγύσεις από την Συμφωνία του Ιουλίου ήρθησαν οι κυρώσεις από πλευρά Ευρωπαϊκής. Χρειάζεται λοιπόν επανάληψη τώρα των ομαλών εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ιράν και του υπόλοιπου κόσμου. Οι ευρωπαϊκέ τράπεζε, ωστόσο, διστάζουν να χρηματοδοτήσουν εμπορικά έργα με το Ιράν, διότι φοβούνται ότι θα του επιβληθούν πρόστιμα από τι ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Έτσι, ενώ υπέγραψε ο Γάλλος, ο Γάλλος πρόεδρος με το Ιράν την πώληση 118 αεροσκαφών Boeing, ε, συγγνώμη, Airbus, αυτό καθυστερεί. Υφιστάμεθα τις επιπτώσεις κυρώσεων που έχουν επιβληθεί ήδη από παλαιών ετών. Αυτά χρειάζεται όμως να γίνουν με γραπτό τρόπο. Να ασαναλάβουν αναλάβουν επιτέλους οι χώρες την ευθύνη τους και ζητήσουν από τη Κεντρική Γαλλική Τράπεζα να χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις γαλλικές για το Ιράν. Ο κ. Μπαλσό, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Ιούλιο 2015 το Ιράν συνήψε συμφωνία με τη διεθνή κοινότητα. Το Ιράν έκανε προσβάσιμο το πυρηνικό του πρόγραμμα σε ελέγχους και καταρχήν ήρθαν οι κυρώσεις. Καταρχήν, διότι ιδίω στον τραπεζικό τομέα οι Ηνωμένε Πολιτείε έκαναν πάντο δυνατό για να διατηρήσουν τις κυρώσεις. Αυτό αντιστατεύεται στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε όμως ομαλές επαφές με το Ιράν. Αυτές τις οποίες προωθούμε. Όμως αυτό δεν αρέσει τις Αμερικανικές αρχές, οι οποίες οφείλουν να άρουν τις κυρώσεις, οφείλουν από την άλλη μεριά να ασκήσουν πίεση στη Σαουδική Αραβία. Διότι η Σαουδική Αραβία κάνει εγκλήματα πολέμου στην Ιεμένη και είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και οδηγεί αυτό βέβαια σε κλιμάκωση των εντάσεων με το Ιράν. Είναι όμως δικό μας συμφέρον να υπάρξει η ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Ευχαριστώ. Η Τόμασίτς. Αυτό τονίζει την λεπτή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παγκόσμιες ε, διπλωματικές, στρατιωτικές και εμπορικές σχέσεις. Είμαστε βασικός εταίρος των ΗΠΑ και γι' αυτό εδώ και πολλά χρόνια χαίρομαι ε, ορισμένων ε, προνομίων. Όμως έχουμε και αρνητικές επιπτώσεις, όπως τώρα με τις επιχειρηματικέ επιχειρηματικές δραστηριότητες ευρωπαϊκών εταιριών στο Ιράν. Ορισμένοι συνάδελφοι χρησιμοποιούν αυτή την ευκαιρία για να αμφισβητήσουν την εταιρική μας σχέση με τη ΣΥΠΑ, αλλά εγώ πιστεύω ότι κάνω λάθος αυτή την περίσταση. Θα πρέπει να οικοδομήσουμε την θέση της Ευρώπης ως ενό ισχυρού ανεξάρτητου ε, φορέα παίκτη που χαίρει τη εμπιστοσύνη των Αμερικανών εταίρων του αλλά και έχει αξιοπιστία προς τους ανατολικούς της ε, εταίρους. Η διασύνδεση της Ευρώπης, της Αμερικής, ε, μάλλον η διασύνδεση των ευρωπαϊκών με τα αμερικανικά συμφέροντα είναι γεγονός, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παίξει πιο ανεξάρτητο ρόλο. Κυρία, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για παράδειγμα του ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Αμερικανική κυβέρνηση μιλούν μεν για το ελεύθερο εμπόριο, αλλά πολύ λίγα πράγματα κάνουν στον χώρο αυτό. Και η Κομισιόν απλώς κάθεται και κοιτάει. Ενώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να φοβούνται την επιβολή προστήμων από τις αμερικανικές αρχές εφόσον προχωρήσουν σε ε, χρηματοδοτήσεις στο Ιράν και επομένως ανακόπτεται οποιαδήποτε δραστηριότητά τους εκεί, σε χαμηλό επίπεδο, τα βλέπουμε τώρα και στο υψηλό επίπεδο. Από το Γενάρη αναμένει η Airbus την άδεια να κάνει ε, πωλήσει στο Ιράν. Και μόλις χθε μάθαμε ότι η Boeing προχωρεί σε πώληση ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν. Πρόκειται για πραγματικό οικονομικό πόλεμο από τις ΗΠΑ, όχι απέναντι στο Ιράν, αλλά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κοιτάζει άπραγη. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριο Φουντούλη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική συνειδητά επιλέγουν να εμποδίζουν τι ευρωπαϊκέ επιχειρηματικέ δραστηριότητε στο Ιράν. Ο λόγο είναι προφανή και φυσικά δεν έχει σε τίποτα να κάνει με δίθεν ανησυχίε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν το βασικότερο που του απασχολεί είναι η προώθηση των αμερικανικών εμπορικών συμφερόντων στη χώρα αυτή. χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση τη airbus που όπω γνωρίζετε έχει κλείσει συμφωνία με την κρατική iran air για την προμήθεια 118 αεροσκαφών από τα τέλη ιανουαρίου. λόγω όμω τη χρήση κάποιων υποσυστημάτων αμερικανική προέλευση απαιτείται έγκριση από την αμερικανική κυβέρνηση για την πώληση των αεροσκαφών η οποία πέντε μήνε μετά δεν έχει δοθεί ακόμα φυσικά η κολυσιεργία αυτή ωφέλισε την αμερικανική boeing που πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε διαπραγματεύσεις με το ιράν για την προμήθεια εκατό δικών της αεροσκαφών. με αυτές τις επιδείξεις συμμαχικής αλληλεγγύης και εμπορικών συναλλαγών όπως τις εννοούν οι αμερικάνοι φροντίζουν να ξεκαθαρίζουν κάθε φορά το ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτή τη συμμαχία. αυτό ας το λάβουν υπόψη τους οι θειασότες των συμφωνιών τύπου ttip για το ποιο θα είναι το μέλλον τη Ένωση, διότι θέματα όπω του ιράν είναι απλά μία εικόνα από το διατλαντικό εμπόριο μέλλον που κάποιοι εδώ πέρα υποστηρίζουν. Ευχαριστώ. Thank you, colleagues. And now... Ευχαριστούμε, συνάδελφοι. Ε, διαδικασία Catch the Eye. Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι εξεδαφικές επιπτώσεις των κυρώσεων του ΙΠΑ τον είπα, κατά το Ιράν εξακολουθούν να δημιουργούν δυσκολίες στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μετά από τις κυρώσεις του 2012 και 2013, οι συνολικές εισαγωγές από το Ιράν μειώθηκαν ε, κατά 38% ε, και οι εξαγωγές κατά 25%. Τώρα οι ΗΠΑ πρέπει να άρουν τα περιοριστικά μέτρα. Αφού το Ιράν ε, είπε ότι θα χρησιμοποιεί την πυρηνική ενέργεια μόνο για πολιτικούς σκοπούς, θα πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για μια πλήρη ένταξη του Ιράν στην διεθνή κοινότητα. Είναι προφανές ότι η επανασύνδεση εμπορικών σχέσεων, επανασύνδεση εμπορικών σχέσεων είναι ένα βασικό στοιχείο για τη σταθεροποίηση της περιοχής και για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Μωράες. Ε, συγγνώμη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι περισσότερε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει δεν αποτολμούν να ανοίξουν δουλειέ με το Ιράν παρά τη συμφωνία του περασμένου χρόνου για το πυρηνικό πρόγραμμα τη Τεχεράνη. Αυτό συμβαίνει επειδή φοβούνται ότι θα του επιβληθούν πρόστιμα από τι Ηνωμένε Πολιτείε για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν που συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δώσει λύση σε αυτό το μείζον ζήτημα που περιορίζει την ανάπτυξη διμερών εμπορικών σχέσεων του Ιράν με κράτη-μέλη τη Ένωση. Η χώρα αυτή των 80 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται σε κατασκευαστικό οργασμό. Στα άμεσα σχέδια είναι κατασκευή 7 αεροδρομίων τα επόμενα χρόνια, ενώ 8 πόλει γνωρίζουν ραγδαία επέκταση. Αυτό το γεγονό ανοίγει τον δρόμο και μπορεί να αποτελέσει ανάσα επιβίωση τόσο για τι κατασκευαστικέ από την Ελλάδα που έχουν πληγεί από τι πολιτικέ τη Τρόικας, καθώ επίση και για ελληνικέ εταιρείε προμήθεια στον χώρο τεχνολογιών εχμής των φαρμάκων των παραφαρμακευτικών προϊόντων αλλά και των ιατρικών ειδών. αναμένουμε κυρία μπιενκόφσκα τη δράση της κομισιόν. ευχαριστώ. Όταν ε, βρέθηκα στο Ιράν, ε, ε, κατά την επίσκεψή μου ήταν σε ισχύ ακόμη οι κυρώσεις, είδα πόσο σημαντικό ήταν για το Ιράν να συνεργαστεί οικονομικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνειδητοποίησα ότι θα ήταν μια ευκαιρία για την Ιρανική οικονομία να προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν πως ακόμη μια φορά παίζουν μαζί μας οι Αμερικανοί έτσι όπως έχει η κατάσταση ε, ε, για η ε, αντιπαράθεση Airbus και Boeing. Παρότι ε, θα το άξιζε η Airbus, νομίζω τελικά η Boeing θα προχωρήσει στις πωλήσει. Ε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε μια μοναδική πολιτική ευκαιρία και θα πρέπει να την ε, αξιοποιήσουμε. από τα μεγαλύτερα σφάλματα της εξωτερικής πολιτικής της ευρωπαϊκής ενώσεως είναι η απόλυτη και ανεξήγητη σύμπλευσή της με εκείνη των ηνωμένων πολιτειών. η αιμονία αυτή έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε χώρες της ευρωπαϊκής ενώσεως και έχει στραφεί πολλές φορές και εναντίον των συμφερόντων της ενώσεως. χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ε, ε, καταστάσεως είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείε των ευρωπαϊκών χωρών που δραστηριοποιούνται στο Ιράν εξαιτία των κυρώσεων που δεν, έχει ακόμη οι δεν έχουν άρει οι Ηνωμένε Πολιτείε για τη χώρα αυτή. Ε, έτσι δημιουργείται μια κατάσταση αθεμίτου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείε και παράλληλα εάν αυτές έχουν συναλλαγές και με τη ηπα κινδυνεύουν να υποστούν κυρώσει, δηλαδή να δεχθούν πρόστιμα αυτό είναι μια απαράδεκτη κατάσταση και πρέπει οπωσδήποτε η ευρωπαϊκή ένωση να απαλλαγεί τάχιστα από αυτή την άτυπη κυδαιμονία για να μπορούν οι ευρωπαίοι επενδυτέ να δραστηριοποιηθούν στην ιρανική αγορά αλλά και στον τομέα τη ενέργεια. Ευχαριστώ. Thank you, uh, ευχαριστώ και τώρα η Σας, ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων ε, που είχαμε και σας ευχαριστώ. Ήταν ξεκάθαρες ε, οι παρεμβάσεις σας. Σίγουρα θα αναλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και συγκεκριμένε περιπτώσεις στις οποίες αναφέρθηκα. Θα επανέλθω σε αυτό στην Airbus και στην Boeing. Εν συντομία βεβαίως. Διαπιστώνουμε πάντως πως ε, το σχέδιο δράση θα πρέπει να λειτουργήσει προς συμφέρον όλων, κυρίως για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και για να ε, ε, ενσωματωθεί και πάλι το Ιράν στην παγκόσμια οικονομία. Θα προσφέρουμε όλη την υποστήριξη που χρειάζεται για προς τις επιχειρήσεις φυσικά θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Για την Airbus μπορώ να σας πω ότι πριν από μήνες υπέγραψε συμφωνία, στα τέλη Ιανουαρίου δηλαδή, ε, όταν ε, ήρθε ο Ιρανός πρόεδρος στη Γαλλία στις 28 Ιανουαρίου για την εξαγωγή αεροσκαφών η Boeing ε, υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης, όχι συμφωνία, πάλι για την εξαγωγή ε, αεροσκαφών, αλλά πολύ πρόσφατα και είναι ε, σε, σχεδόν στην ίδια κατάσταση αυτές οι δύο εταιρείες. Ε, η διαφορά είναι ότι είναι συμφωνία για την Airbus και μνημόνιο για την Boeing. Ξέρουμε Φυσικά ότι θα πρέπει να συνεχίσουν όλες οι πλευρές τις προσπάθειές τους. Θα διαβιβάσω τα σχόλιά σας ε, στην κυρία Μογκερίνη και σας ευχαριστώ που γράψατε το σημείο στην μερίσια διάταξη. Ελπίζω να μας απασχολήσει και στο μέλλον το θέμα, διότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την ευρωπαϊκή οικονομία.